Koleżanki i koledzy, συνάδελφοι, ξεκινά η συνεδρίασή μας και έχω κάποιες ανακοινώσεις να κάνω. Καταρχάς ανακοινώνω τη συνέχιση της διακοπής σας συνόδου που είχε διακοπή στις 17 Φεβρουαρίου. Τα πρακτικά της προηγούμενης συνόδου είναι στη διάθεσή σας. Υπάρχουν σχόλια. Δεν νομίζω να υπάρχουν σχόλια. Άρα θεωρούνται τα πρακτικά ως ε, εγκεκριμένα. Θα ήθελα να σας δώσω, να κάνω τις ανακοινώσεις, σας δώσω κάποιες πληροφορίες. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι η γραπτή δήλωση 89 κάθετος 2010 έχει συλλέξει τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών και γι' αυτό έγινε κείμενο υιοθετημένο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτή η δήλωση εντάσσεται στη μονομερή επαναφορά των απαιτήσεων ε, θεωρήσεων από τον Καναδά για τους Τσέχους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναμένει το ε, το Συμβούλιο να λάβει μέτρα όσον αφορά ε, το Καναδά, ούτω ώστε να καταργηθεί αυτή η απέτηση για θεώρηση ταξιδίων, θεώρηση διαβατηρίων για τους τσέχου υπηκόους. Είμαστε αλληλέγγυοι με τους πολίτες της Τσεχική δημοκρατίας που όπω οι άλλοι ε, υπήκοοι των κρατών των άλλων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα έπρεπε να μπορούν να μπαίνουν στον Καναδά χωρίς βίζα. Μετά, Δήλωση 2. Στις 11 Μαρτίου για 7η φορά θα γιορτάσουμε την Ευρωπαϊκή ημέρα των θυμάτων της τρομοκρατίας. Αυτή την ημέρα, το 2004, έγιναν οι βομβιστικές επιθέσεις στη Μαδρίτη και σκότωσαν περίπου 200 ανθρώπους. Και αργότερα μετά από 6 μήνες στο Λονδίνο σκοτώθηκαν 52 άνθρωποι. Δεν δικαιολογείται που δεν είναι η τρομοκρατία καμία τρομοκρατική επίθεση, κανένας τρομοκράτης δεν θα μπορέσουν να αποδυναμώσουν το πνεύμα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και της ε, δημοκρατίας. Και τώρα τρίτη πληροφορία. Έχουμε λάβει κάποιες πληροφορίες που δημιουργούν ανησυχίες όσον αφορά την επαναφορά της θανατικής ποινής στην Ταϊβάν για πέντε άτομα που περιμένουν εκτέλεση. Η επαναφορά λοιπόν της θανατικής ποινή το 2010 ε, ε, κατήργησε το de facto moratorium που υπήρχε από το 2006. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιο συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν κατά της θανατικής ποινή και γι' αυτό ζητούμε από τις αρχές της Ταϊβάν να επανεισάγουν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 Όπως ε, βλέπετε και ακούτε, αυτές οι ανακοινώσεις ισχύουν εξίσου για το 2012 και το 2013. Είναι η ίδια διαδικασία. Τώρα έχω την επόμενη ανακοίνωση. Ο κ. Τζο Higgins και ο κ. Άλαν Κέβιν με ενημέρωσαν ε, γραπτός για την εκπνοή της ε, θητείας τους ως ευρωβουλευτές λόγω του ότι εξελέγησαν στο Ιρλανδικό Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποδέχεται αυτές τις πληροφορίες και σύμφωνα με την αντίστοιχο, το αντίστοιχο άρθρο του εσωτερικού κανονισμού που αφορά την εκλογή Ευρωβουλευτού ε, σε Εθνικό Κοινοβούλιο στις εκλογές δηλώνει ότι αυτές οι δύο έδρες είναι κενές από τις 25 Φεβρουαρίου ε, τους έτους. Και τελευταία ανακοίνωση η υπογραφή των νομικών πράξεων ε, γίνεται, λαμβάνει χώρα μέσα της κανονικής, της συνηθισμένης διαδικασίας. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου και τη Δευτέρα και εγώ θα υπογράψουμε τέσσερις πράξεις δυνάμει το άρθρο 74 ε, του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σημειώνω ότι θα δημοσιευτούν οι πράξεις στα πρακτικά της ε, τριχούσης συνόδου θα δημοσιευθούν στα πρακτικά. Νομοθετικές πράξεις θα δημοσιευθούν αυτές στα πρακτικά. Και πάμε στον καθορισμό του προγράμματος αυτής της εβδομάδας, της συνόδου μας αυτής. Το τελικό σχέδιο προγράμματος υθετήθηκε στις 3 Μαρτίου από τη διάσκεψη των Προέδρων σύμφωνα με το άρθρο 137 του εσωτερικού κανονισμού και σας έχει δοθεί αυτό το σχέδιο του προγράμματος. Λοιπόν, καθημερινά θα καθορίζουμε την ημερήσια διάταξη. Τη Δευτέρα, λοιπόν, δεν έχουμε καμία αλλαγή όσον αφορά την αρχική μας πρόταση. Την Τρίτη, προσέξτε, την Τρίτη έχει γίνει μια αλλαγή. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων υιοθέτησε έκθεση του κ. Σπερόνιου όσον αφορά την άρση ασυλίας του κυρίου Έρμαρ Μπροκ. Σύμφωνα με τις πολιτικές ομάδες και δυνάμει του άρθρου 138, αυτή η έκθεση θα συμπεριληφθεί στην ψηφοφορία αύριο. Είναι η κανονική συνηθισμένη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 138 του εσωτερικού κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Την Τετάρτη και την Πέμπτη δεν έχουμε κάποιες προτάσεις για κάποιες αλλαγές σε σχέση με το πρωταθέν πρόγραμμα, οπότε μπορούμε να θεωρήσουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα ως εγκεκριμένο και μπορούμε να προχωρήσουμε στην πρώτη έκθεση. Συντάκτης είναι ο η κυρία Άννη υποδηματάει η συνάδελφός μας, και ενωτόμα χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος Οντί κάτι θέλει να πει, έχετε το λόγο. Θα ήθελα να μιλήσω, ο κύριο Οντί, θα να μιλήσω δυνάμει το άρθρο 16 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτή την εβδομάδα, κατόπιν πρωτοβουλίας του αρχηγού του κράτους, το οποίο νίκο του Νικολά Σαρκοζή, που ζητά ε, ε, να γίνει έκτακτο Συμβούλιο Ευρωπαϊκό την Παρασκευή να συνεδριάσει. Ήθιστε